Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, αρχίζει η συνεδρίαση. Καλή σας μέρα. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Μακάρθη με θέμα εφαρμογή στα κράτη-μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια. Θα ξεκινήσουμε την συζήτηση με την εισηγήτρια. Κυρία Μακάρθη, θα πάρετε το λόγο για τέσσερα λεπτά σας παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κυρία εισηγήτρια. Ε, Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι έχω έξι λεπτά, αλλά θα τα καταφέρω στα τέσσερα λεπτά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους